η συνεδρίαση. Για διαδικαστικό, ο κύριος Φέρμ. στην, στο κάθισμα 235. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της παρούσας περίοδου συνόδου ρωτήσατε τον αυστριακό συνάδελφό μου Φριντ σχετικά με τα νέα μέλη. Δεχτήκατε μάλλον μια ερώτηση δεχθήκατε μια ερώτηση από τον συναδελφό μου για σχετικά με του νέου ευρωβουλευτέ και είπατε ότι τώρα την πρωτοβουλία κινήσεων έχει το Συμβούλιο. Συμφωνώ, αλλά δεν είμαι βέβαιο όσον αφορά το ενδεχόμενο καθεστώ παρατηρητών πριν να ε, γίνουν πλήρη μέλη. Έχουμε και την έκθεση David Martin καθώ και, και τον κανονισμό μα. Δηλαδή έχουμε την ελευθερία να επιτρέψουμε στα πρόσωπα αυτά να αρχίσουν να συμμετέχουν ω παρατηρητέ, αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί. Εμεί ω Κοινοβούλιο μπορούμε να αποφασίσουμε για του όρου και συνθήκε υπό του οποίου μπορούν να συμμετάσχουν ως παρατηρητέ. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, συζητήστε το με τον εισηγητή κύριο Μάρτιν ώστε να υπάρξει μια λύση το δυνατόν συντομότερο. Θα ήταν πραγματικά παράλογο τα νέα μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί όπου η εκλογή τους έχει κυρωθεί από τις ε, αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας τους να μην μπορούν να αρχίσουν το έργο τους εδώ για μήνες ολόκληρους. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Όπως είπα και πριν, έθεσα ερώτηση στο Συμβούλιο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών, της δικής μας δηλαδή, θα πρέπει να λάβει το θέμα υπόψη του και να το μελετήσει. Δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τον αριθμό των νέων ε, βουλευτών και από ποια χώρα θα προέρχεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Δεν είναι τελική απόφαση ακόμα, δεν έχει ακόμη λάβει τελική μορφή. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να υποδεχθούμε εδώ παρατηρητές εφόσον δεν έχουμε ακόμη την τελική απόφαση σχετικά με τον αριθμό τους και τον αριθμό αναχώρα. Θα πρέπει πάνω λοιπόν να περιμένουμε λίγο. Βέβαια το μελετούμε, το σκεπτόμαστε διαρκώς και πολύ εντατικά. Η κυρία Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να διευκρινίσει το θέμα. Δεν το θεωρώ αδύνατο. Από, την, από τη σκοπιά της ομάδας μου για την συζήτηση για την Γαλλία θεωρώ ότι είναι αφόρητο ή θα ήταν αφόρητο εάν οι παρατηρητές με οποιοδήποτε καθεστώς εξακολουθούν ταυτόχρονα να είναι βουλευτές των εθνικών βουλών. Εμείς θεωρούμε ότι όσοι προσέλθουν εδώ ως παρατηρητές θα πρέπει να παρετηθούν από τις εθνικές τους βουλευτικές έδρες. Ο πρόεδρος σας ευχαριστώ. Άλλο διαδικαστικό. Ο κ. Όντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα απολογισμό της Ιουδικής Προεδρίας που ήταν ε, αποτελεσματική και ε, χρήσιμη. Όμως πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 10 και 11 Δεκεμβρίου. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του ε, Πρόεδρου της Κομισιόν ως θεματοφύλακα της συνθήκης το άρθρο 15.6 της συνθήκης που προβλέπει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάσει μια έκθεση μετά από κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Βαν Ρομπόη δεν θα είναι εδώ. Το θεωρώ αυτό ατυχές και λυπηρό. Έχει εκλεγεί από την 1η Δεκεμβρίου. Έχει ε, εντατικές διπλωματικές επαφές ε, και ε, διεργασίες να αναλάβει και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ευτυχές ως πρώτη πολιτική χειρονομία να έρθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της 10 η και 11 η Δεκεμβρίου. Ε, dziękuję Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε μάλλον, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας εξηγήσω. <clears throat> Υπήρξε συμφωνία που συνήθη μεταξύ των ε, Πρόεδρων κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του κυρίου Βαν Ρομπόη και της παρούσας Προεδρίας του Συμβουλίου, του Πρωθυπουργού κ. Ράινφελτ δηλαδή, σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, για, την, για τον τελευταίο μήνα του παρόντος έτους, θα ισχύσει το παλαιό καθεστώς. Δηλαδή, ο κ. Βαν Ρόμποϊ θα αναλάβει τα καθήκοντά του επισήμως από 1η Ιανουαρίου 2010. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα με την ευκαιρία ο κύριος Οντή. Όχι, Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατό να το δεχτώ αυτό. Είναι μια συνθήκη που έχει επικυρωθεί από του λαού. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να μα παρουσιάσει τον απολογισμό αυτών των συνεδριάσεων. Κύριε συνάδελφε, αυτό αποτελεί μέρο και αποφάσεω του Κοινοβουλίου, δηλαδή και δική σα, που έχει σχέση με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο. Έχουμε και εμείς λάβει δηλαδή την απόφαση αυτή ως Κοινοβούλιο για το ποιον προσκαλούμε και με ποια σειρά. Αυτό το κάνουμε στα πλαίσια της διαθεσμικής μας συνεργασίας. Ίσως λοιπόν είναι πρόωρα τα σχόλια αυτά και εν πάση περιπτώσει συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι είναι ακόμα, όπως είπα, πρόωρο να το συζητήσουμε περισσότερο. Προσπαθούμε πάντως να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ Προεδρίας, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα προκειμένο του κ. Βαν Ρόμποη. Όπως ξέρετε, η Προεδρία θα αλλάξει, αλλά ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει στην θέση του και ε, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση <clears throat> η οποία ασκεί την ε, Προεδρία. Δική μας είναι η απόφαση για τον οποίο θα προσκαλέσουμε. Αλλά αγαπητέ κύριε συνάδελφε, βρίσκω ότι είναι ακόμη πρόωρο να ε, λάβουμε άλλη δράση επί του προκειμένου. Έχουμε τώρα τον Σουηδό Πρωθυπουργό, ο οποίο θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα του εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Ο κ. Βαν Ρομπόη δεν ανεμίχθη σε αυτή την Προεδρία εφόσον ε, διορίστηκε μόλις προ δύο εβδομάδων. Ε, συμφωνείτε κύριε συνάδελφε. Καλώ. Καλώς, καλωσορίζω ιδιαίτερα θερμά τον Πρωθυπουργό κ. Ράινφελτ μετά από ένα σχεδόν εξάμεινο ε, προεδρίας, η οποία λήγει βέβαια στις 31 Δεκεμβρίου.